Έτσι ε, επιβεβαιώνουμε την εντολή. Η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων ε, ε, προτείνει μια ερμηνεία σχετικά με τις αποστολές ενημέρωσης για εξέταση αναφορών. Υπάρχει το κείμενο της ερμηνείας στο Seance Undirect» από την ομάδα των Πρασίνων και το ΕΛΚ ε,